από τις 9 ως τις 13.30, από τις 15 ως τις 20.30, από τις 21 ως τις 24. Η μερίσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνεδρίαση έριξε.